Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι για μια φορά ε, ομοφωνούμε εδώ για την τράπεζα. Ευχαριστούμε κύριε Σμίτ, εδώ ολοκληρώνει τη συζήτηση και αύριο στις 11.30 θα γίνει ψηφοφορία για το κείμενο αυτό. Και τώρα πάμε στην έκθεση σκήνου που αφορά τα συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων. Και δίνω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Σάντσες Πρεσέδο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αντικαταστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πίτερ Σκίνερ, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι παρόν και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω σε αυτή τη συζήτηση που τόσο θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτήν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα και στο όνομά του να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για το θαυμάσιο πλαίσιο συνεργασίας που δημιούργησαν μαζί του για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Η έκθεση για τα συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι ασφαλισμένοι θα, είναι, θα έχουν κάποια εγγύηση έναντι μιας ενδεχόμενης πτώχευσης της εταιρείας ασφάλισης και επομένως διατήρησης των ωφελημάτων που προκύπτουν από το ασφαλιστικό του συμβόλαιο. Τα συστήματα εγγύηση που ισχύουν αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν διαφορετικέ πτυχέ και αντανακλούν τις, ε, τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εθνικών αγορών. Η έκθεση αυτή υποστηρίζει την επίτευξη ενό ελάχιστου επίπεδου εναρμόνισης που εξασφαλίζει κάποιο κοινό παρανομαστή σε όλα αυτά τα συστήματα, τα διαφορετικά που υπάρχουν στα κάτι μέλη. Ζητά επιπλέον αυτή η έκθεση να προτείνει, να προτείνει η Κομισιόν μια οδηγία για διαμεθοριακή εναρμόνιση που να εξασφαλίζει ένα συνεκτικό επίπεδο προστασία των καταναλωτών και ασφαλισμένων για όλα τα προϊόντα στον ασφαλιστικό τομέα. Επίση, ζητά από την Κομισιόν να προχωρήσει σε εκθέσει αντικτύπου που να είναι λεπτομεριακές και δημόσιες διαβουλεύσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών ασφαλιστικών συμβολέων, ώστε να υπάρχει ένα ισόπεδο γήπεδο μέσα, μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ζητά επίση η έκθεση από την Κομισιόν να θεσπίσει ένα ενιαίο υπόδειγμα για τη χρηματοδότηση από τις εταιρείες ασφαλίσεων για τα συστήματα προστασίας των ασφαλισμένων σε περίπτωση πτώχευσης των εταιρεών. Εμείς χαιρετίζουμε θετικά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο οδηγίε για τα θέματα αυτά. Θα ήθελε ο κύριο Σκίνερ περαιτέρω να διαβιβάσει σε όλους σα την προσήλωσή του στο να συνεχίσει σε πνεύμα συνεργασία να συνεχίσουν οι προσπάθειες στα διάφορα άλλα νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό σύστημα και τα οποία συζητούνται τώρα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Σάντσεφ Πρεσέδο. Η κυρία Φόρδ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Παρακαλώ διαβάστε τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή και ξέρω πως θέλετε να υπάρξει ένα συνεκτικό διασυνοριακό πλαίσιο για την ασφάλιση αυτή και σεβασμό βεβαίως πάντα της επικουρικότητας. Δεν θα ψηφίσω όμω αυτή την έκθεση γιατί το κόστο ασφάλιση ανεβαίνει σε πολλέ χώρε και σε πολλού ε, κλάδου. Σήμερα ασφαλιστικέ εταιρείε ε, αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού, υψηλότερε απαιτήσει φερεγγιότητα, αλλά είναι πιο εκτεθειμένε στην απάτη και βεβαίω υπάρχουν και υπερβολικέ απαιτήσει ει βάρο του. Και όλα αυτά πριν η Επίτροπο Ρέντινγκ ξεκίνησε να μιλάει για τι γυναίκε οδηγού κινδυνεύουμε η ασφάλεια να γίνει πάρα πολύ ακριβή για όσους έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και πολύ συχνά η Κομισιόν καταθέτει νομοθετήματα τα οποία προσθέτουν κόστος χωρίς να προσθέτουν όφελος. Θα αναμείνω να δω ποιες είναι οι προτάσεις της ε, Κομισιόν πριν κρίνω. Κατ' ουσίαν, ποιο είναι το όφελος του να προσφέρουμε περαιτέρω προστασία των καταναλωτών εάν μείνουν πίσω καταναλωτές οι οποίοι δεν θα μπορούν πλέον να αγοράσουν αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η οικονομική κρίση έδειξε πως η εμπιστοσύνη των καναλτών εξασθενεί και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν και ε, πολύ λίγες αποζημιώσεις ε, στην περίπτωση κάποιου ασφαλισμένος. Θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν ε, αυτές οι ασφαλίες στην περίπτωση, οι αντασφαλίες στην περίπτωση στην οποία χρεοκοπήσει η ασφαλιστική εταιρεία. Όμως ε, οι αντασφαλιστικές εταιρείε διαφέρουν ε, όσον αφορά την κάλυψη των καταναλωτών και Υπάρχουν και διαφορετικά κριτήρια και αν θέλει βεβαίως κανείς να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών, νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα προστασίας των καταναλωτών. Οπότε, ειλικρινά, ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει πως ε, ό,τι και αν είναι ε, ασφαλισμένος και υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης 100% εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει στους καταναλωτές μια προστασία στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία απαιτούνται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση, ο τομέας αυτός θα οδηγεί όλο και περισσότερο σε στρεβλώσεις σε διαμεθοριακό επίπεδο και θα μειώνει το επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Η Ρουμανία μεταξύ των 11 κρατών μελών που έχουν ένα γενικευμένο σύστημα εγγυήσεων των ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι το πάνω από το, μεγαλύ... πάνω ίμιση της αγοράς ασφαλίσεων στην Ευρώπη δεν έχει συστήματα προστασίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει πλήρω την εγγύηση των ασφαλίσεων και να μπορεί να δώσει ε, αποζημιώσει στου ασφαλισμένου σε περίπτωση πτωχεύση τη επιχείρηση που του ασφαλίζει. Είναι απαραίτητο όμω το μοντέλο χρηματοδότηση για το Ταμείο Αυτό Εγγύσεων να σέβεται την αρχή τη επικουρικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Μπασέσου. Κύριο Σκέλ. Χαιρετίζουμε στην έκθεση Σκίνερ. Στους καιρούς που είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση ασφάλειας και έχουμε ένα παράδοξο και στη δική μου χώρα. Πέφτουν οι μισθοί. Παρ' όλα αυτά τα ασφάλιστρα έχουν εκτιναχθεί. Για όλες τις ασφαλίσεις λέω. Κυρίως για την ασφάλιση υγείας. Δεν μπορεί να καλυφθεί όλος ο κόσμος. Δεν είναι ικανοποιητικό Είχαμε πλημμύρε, εξαπλασιάστηκαν εκεί τα ασφάλιστρα. Και πάρα πολλέ φορέ οι όροι στα ψηλά γράμματα των ασφαλιστερίων είναι ναρκοπέδι. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δίκαιε συνδικέ τόσο ώστε να ότι θα υπάρχει αυθεντική ασφάλιση των καταναλωτών. Και όντω να ασφαλίζονται ανάλογα με αυτά τα οποία καταβάλουν. Ευχαριστούμε κύριο Πάσκα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, το 2013 πρόκειται η οδηγία για την πτώχευση θα τεθεί σε ισχύ και θα επηρεάσει την αγορά. Όπως έχει σήμερα η νομοθεσία, δεν καλύπτονται οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εναρμονίσει τις σχετικές διατάξεις μέσω της οδηγίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο και τι να κάνουμε, ας γίνει η εναρμόνιση με τον ελάχιστο κοινό προνομαστή. Και ο Γιάννης Επικουρικότητας βέβαια πρέπει να χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να υπάρχει όσο είναι μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη από την ρύθμιση. Βέβαια πάντοτε υπάρχει η αρχή της ε, χώρας της έδρας της εταιρεία. Πρέπει να επομένως προς ε, κατοχήρωση των εγγύσεων. Κάτσε τη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το... Η διαφορά στα συστήματα εγγυήσεων των ασφαλίσεων είναι προϊόν των διαφορετικών καταστάσεων που ισχύουν στις χώρες μέλη μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει σε ποιο σύστημα, ποιο σύστημα τον καλύπτει. Τα συστήματα λοιπόν εγγυήσεων των ασφαλίσεων θα πρέπει να δίδουν το ίδιο επίπεδο προστασία σε όλους τους καταναλωτές, αποζημιώσεις για ζημίες που υφίστανται και αυτό να περιλαμβάνει την ε, περίπτωση αφαιρεγγιότητος του Ιδρύματος του Πιστοτικού του Ασφαλιστικού, το οποίο παρέχει την προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα προστασίας των καταθέσεων και να υπάρξει μεγαλύτερη ομοιογένεια στην αγορά <clears throat> ασφαλίσεων. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής θα την χάνει ίσης προστασίας ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται, ανεξάρτητα από τους κινδύνους που καλύπτονται από το Ασφαλιστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ρέν κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σκίνερ ε, και τον κύριο Σάντσε Πρεσέλα που τον αντικαθιστά και την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων για τα ζητήματα εγγύησης των ασφαλίσεων. Πρόκειται λοιπόν για μια απόπειρα να ξεπεράσουμε το κατακαιρματισμένο πλαίσιο που υπάρχει μέσω της ελάχιστης εναρμόνισης. Σκοπεύουμε να καταθέσουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του 2012 πρόταση οδηγίας. Υποθέτω πως συμφωνούμε όλοι με αρκετά από αυτά τα οποία ακούστηκαν όπως παραδείγματο χάρη την ε, αρχή του Κυριού και την δυνατότητα και τη έδρα τη ε, εταιρεία. Και βεβαίως ε, πρέπει να υπενθυμίσω πως ε, η θέση της Κομισιόν δεν συμφωνεί πλήρως με την έκθεση όπως αυτή υποβλήθηκε σήμερα. Η θέση μας στην η λευκή βίβλο ήταν πώ θα έπρεπε να καλύπτει ασφαλή ζωή και μη. Όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης, η Λευκή Βίβλος όριζε πως θα έπρεπε να οριστεί ένα κατάλληλο επίπεδο στόχου χρηματοδότησης σε μια λογική περίοδο και εάν η χρηματοδότηση τώρα θα πρέπει να είναι εξάντε ή εξπόστ στη Λευκή Βίβλο η θέση μας ήταν πως το σχέδιο αυτό σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να χρηματοδοτείται ως ένα βαθμό με συνεισφορές εξάντε από τις ασφαλιστικές εταιρείε. Όμως η Κομισιόν δεν απέκλεισε στην περίπτωση έλλειψης πόρων να συμπληρωθούν τα κεφάλαια με χρηματοδότηση ex post. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η έκθεση του κυρίου Σκίνερ έρχεται σε μια σημαντική στιγμή. Προετοιμαζόμαστε για ένα Ευρωπαϊκό Καθεστώ Εγγύηση των ασφαλιών και θεωρούμε πως δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στο μέλλον να βρούμε περιθώριο συνεννόησης για το ε, Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Και μας ενθαρρύνει βεβαίω η διάθεση την οποία δείξατε και η έκθεση αυτή, η ενισχύ αυτή τη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11 και 30 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τώρα την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας μετά τη θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας.